Ε, Καλό απόγευμα σε όλους. Καλωσορίσατε στην Στρογγύλη Τράπεζα Υπαριθμών 2 στα πλαίσια της ε, διάσκεψης υψηλού επίπεδου. Λέγομαι Τόμας Τομπέ. Είμαι πρόεδρος ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι στη Σουηδία, την πατρίδα μου και από εδώ σας μιλώ. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε αυτήν την ε, διάσκεψη με συμμετοχή από απόσταση λόγω της ε, πανδημίας ε, COVID. Πάντως, να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που να συμπροεδρεύσω με την ε, Σλοβενή συνάδελφό μου αυτήν την στρογγυλή τράπεζα που ε, θα είναι αφιερωμένη στην εξωτερική διάσταση της, ε, του ασύλου και της μετανάστευσης υπό τον τίτλο Shaping Partnerships with Third Countries. Να σας πω ότι έχουμε μετάφρα διερμηνία σε 7 γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, φινλανδικά, ελληνικά και σλοβενικά. Μπορείτε να ακούτε και να μιλάτε ελληνικά από πλευράς ε, του Κοινοβουλίου ε, αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών βρίσκεται πραγματικά ε, στην καρδιά, στο επίκεντρο της σημερινής διάσκεψης υψηλού επίπεδου για την μετανάστευση και το άσυλο. Επομένως είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων προς τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν ήδη καταγραφεί να συμμετάσχουν στη στρογγυλή τράπεζα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη Γερμανική Βουλή Bundestag που είναι συνδιοργανωτή αυτής της σημερινής μας ε, συνεδρίασης. Επίσης, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μα, Μαρία Ρενά, ε, τον ε, πρόεδρο του, της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής, Υποεπιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που θα έχουμε μαζί μας την Επίτροπο Ουπ την Επίτροπο κυρία Μύρα Ελφάντη, για την Αφρικανική Ένωση και επίσης τον κύριο Νίκολα Μπέι από το, ε, τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης Επίσης, ε, ε, τέλος, ε, να ευχαριστήσω ιδιαίτερο την συμπρόεδρό μου, κυρία Μόνικα Γκρεγκόρτσιτς, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Σλοβενικής Βουλής. Αγαπητή κυρία Γκρεγκόρτσιτς, θα συμπροεδρεύσουμε αυτήν την στρογγυλή τράπεζα και πραγματικά θα έχουμε μια πολύ ωραία χορογραφία μεταξύ μας. Το 2015 ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και πραγματικά μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική για την πολιτική ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί αφορά στην ουσία τις ε, αρχές της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον ε, Σεπτέμβριο ξεκίνησε και η διαδικασία για μια νέα δέσμη όσον αφορά την ε, ε, μετανάστευση και το άσυλο και προτείνει μια ολιστική συνολική προσέγγιση των θεμάτων αυτών. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την εξωτερική διάσταση των θεμάτων. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτά να αντιμετωπιστούν σε πλαίσιο συνεργασίας και κοινή προσπάθειας. Ε, πρέπει να υπάρξει μια καλή οικοδόμηση ικανοτήτων έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά και τις ανάγκες των μεταναστών προσφύγων. Θα πρέπει επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις ε, βασικές αιτίε της μετανάστευση η νέα δέσμη ε, για την μετανάστευση μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναρχίσουμε με νέο τρόπο και εξ αρχής ε, και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις ε, που παρουσιάζει το θέμα της μετανάστευσης σήμερα. Η αλληλεγγύη βεβαίως βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της δέσμης και είναι πάρα πολύ σημαντική για να λειτουργήσει καλά το σύστημα της μετανάστευσης και του ασύλου. Η Επίτροπος κυρία Λάινεν θα ε, μπορέσει να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ε, ε, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο η κάθε χώρα μπορεί να συμβάλλει έτσι ώστε συνολικά να αντιμετωπιστεί το θέμα της μετανάστευσης που βεβαίως είναι στενά συνδεδεμένο με το θέμα της ένδυας, της φτώχειας Κυρίες και κύριοι, η ανάγκη αλληλεγγύης προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι πολύ σημαντικό, αλλά βεβαίως ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να έχουμε την διαδικασία εξωτερικής βοήθειας, αλλά με ταυτόχρονο σεβασμό των ε, δικαιωμάτων των αρχών μας, επί των οποίων βασιζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην οικονομική ε, και κοινωνική ανάπτυξη των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των χωρών της εταιρικής σχέσης. Μαζί μπορούμε να παίξουμε σημαντικότερο ρόλο. Τώρα θα δώσω το λόγο στην συμπρόεδρό μου, την κυρία Μόνικα Γκρεγκόρτσιτς, από την Εθνική Βουλή της Σλοβενίας. Παρακαλώ κυρία Γκρεγκόρτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Τομπέ. Είναι και για μένα ιδιαίτερη τιμή να συμπροεδρεύουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και λοιποί αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα, στα σλοβενικά. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που έχουμε καταφέρει να ε, υλοποιήσουμε αυτή την, ε, ε, αυτή την ιδέα μάλλον που είχαμε για την διοργάνωση ενός πάνελ υψηλού επίπεδου και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και επίσης την Γερμανική, το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Bundestag, για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Πρώτη φορά διοργανώνεται μια τέτοια συζήτηση. Και Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις εισαγωγικές για το θέμα μας. Στο ζήτημα της μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιορίζεται στην προστασία των εξωτερικών της συνόρων. Θα πρέπει να συνεργάζεται με χώρες κλειδιά, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης. Υπό αυτήν την έννοια θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις τρίτες χώρες, είτε πρόκειται για χώρες προέλευσης, είτε πρόκειται για χώρες διέλευσης. Είναι κρίσιμο αυτό για να υπάρχει μια ουσιαστική ε, και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αυτή η εταιρική σχέση θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τρίτη χώρα. Οι σχέσεις αυτές θα πρέπει όχι απλώς να μας επιτρέπουν να καταπολεμούμε την εμπορία ανθρώπων ή να βοηθούμε εκείνες τις χώρες που ε, φιλοξενούν πρόσφυγες, αλλά ταυτόχρονα να μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τα γενεσιουργά αίτια ε, και τα προβλήματα στις χώρες από τις οποίες έρχονται οι μετανάστες. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές διεθνώς. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ρωτηθούμε εάν αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια ε, είναι σωστά στοχευμένη και αν πράγματι μειώνει την ανάγκη των ανθρώπων να μεταναστεύσουν. Κατά την άποψή μου χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα, των κρατών μελών της για να έχουμε καλύτερη στόχευση της αναπτυξιακής αυτής βοήθειας, να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες διαβίωσης στις τρίτες χώρες και να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι η μετανάστευση είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χαίρομαι που έχουμε στην συζήτησή μας σήμερα και οργανισμούς εκτός Ευρω... Ευρώπης. Ε, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να έχουν συντονισμένη ανταπόκριση σε αυτή την πρόκληση, αλλά για να βρούμε μια πραγματική λύση χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία, ε, πολυμερής. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία με τους συναφείς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνέ επίπεδο, όπω η Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, διάγουμε δύσκολους και καιρούς και θα πρέπει να επιδείξουμε φιλοδοξία, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και ρεαλιστές. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την ευημερία και τη σταθερότητα παγκοσμίω με αυτέ τι σκέψει θα ήθελα να σα παρουσιάσω τώρα τον τρόπο που θα οργανώσουμε τη σημερινή μα συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις από τους δύο προσκεκλημένους μας υψηλού επίπεδου, δηλαδή την Επίτροπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επίτροπο της Αφρικανικής Ένωσης. Μετά θα συντονίσει ο κύριος Τομπέ μια συζήτηση ε, και ένα πρώτο, το πρώτο σκέλος της συζήτησης με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ θα προεδρεύσω στο δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτά από την πλευρά μου. Θα ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Τομπέ. Ε, μάλλον τέλος θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Τομπέ ε, για να ολοκληρώσουμε το πάνελ. Ε, θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας παρουσιάσω τους δύο προσκεκλημένους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Αφρικανική Επιτροπή. Τελεί τιμή για μένα να, προσ... να ε, καλωσορίζω μάλλον εδώ την κυρία Γιούτα Ουτπιλάινεν, ε, ε, Επίτροπο Αρμόδια για τις Διεθνείς Συνεργασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Αμύρα Ελφαντήλ, τον κύριο μάλλον Αμύρα Ελφαντήλ, από την Αφρικανική Ένωση, Επίτροπο για τις Κοινωνικές Υποθέσεις. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, αγαπητοί Επίτροπη, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Επίτροπο Ούρπι για 7 λεπτά. Commissioner Ulpilainen, are you... Μας ακούτε κυρία Ulpilainen. Commissioner, we Μπορούμε να δούμε την εικόνα από το γραφείο της Επιτρόπου, αλλά δεν σας ακούμε. Ε, θα προσπαθήσουμε να ε, βελτιώσουμε τη σύνδεση. Ένα λεπτό. we cannot hear you. Συνεχίζουμε να μην μπορούμε να σας ακούμε. Να σας ζητήσω το εξής. Μπορείτε να αποσυνδέσετε τα ακουστικά με το μικρόφωνο που χρησιμοποιείτε για να δούμε αν θα δουλέψει η συσκευή σας χωρίς. still have no sound on... Όχι, ακόμα δεν έχουμε ηχό, δυστυχώ. Θα επικοινωνήσει κάποιο από του τεχνικού μα με το γραφείο σα για να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν, δεν, δεν φτάνει ο ήχο σε εμά. Um, yes, we will try to... Ε, ε ναι, λέει η κυρία Γκρεγκόρτσιτ, ε, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Εν τω μεταξύ όμω, προτείνω να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μα και θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω την Επίτροπο κυρία Αμύρα Ελφαντήλ, και να της δώσω τον λόγο για 7 λεπτά. Κυρία Αλμύρα, Αμύρα Ελφαντήλ. Μας ακούτε κυρία Ελφαντήλ. Hello? Hello? Yes, we can see you and hear you. You can see me and hear me because I had to use the headphones to hear you. Λοιπόν, μια και λύσαμε τα τεχνικά προβλήματα, να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ελφαντήλ. Κύριε Τόμας Τομπέ, ε, ε, ε κυρία Μόνικα ε, Γκρέγκορτσιτς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την ε, ε, Σλοβενική Βουλή, Βουλή τον κύριο Νικόλα Μπέι από το Συμβούλιο Προσφύγων της ε, ε, Δανίας. Ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την, και όλους όσοι μας έδωσαν την ευκαιρία αυτή να είμαστε εδώ και να συμμετάσχουμε σε αυτήν την σημαντική διακοινοβουλευτική υψηλού επίπεδου συνάντηση με θέμα την ε, μετανάστευση και το άσυλο λόγω της ιστορίας ε, και λόγω του παρελθόντος, του παρόντος αλλά και του κοινού μέλλοντος ε, η Αφρικανική Ένωση ε, θέλει συνεργασία όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις δημοτικές αξίες. Διεθνείς συμφωνίες έχουν υπάρξει μεταξύ των αντιστοίχων ενώσεών μας. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο στενός γείτονας, κοντινός γείτονας, είναι και στενός συνεργάτης. οι δύο ήπειροι μας έχουν συνεργαστεί τις τελευταίες ε, δεκαετίες σε θέματα ενέργειας, σε θέματα μετανάστευσης, θέματα κλιματικής αλλαγής, κινητικότητας, καθώς επίσης και άλλα πολλά θέματα. Η εταιρική ε, σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αφρικής ε, θέλει να δημιουργήσει μια καλή οικονομική συνεργασία αλλά και βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη. Αυτού του είδους οι διασκέψεις βοηθούν την ανάπτυξη διαλόγου και την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου έτσι ώστε να ενδυναμωθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο υπήρων για θέματα κινητικότητας και μετανάστευσης. Ο διάλογος επίσης έχει στόχο την επιτάχυνση 7 προτεραιοτήτων που συμπεριλαμβάνουν τα εμβάσματα και τις αδυνατότητες επενδύσεων καθώς επίσης και την ανταλλαγή εμπειριών και ε, ε, θεμάτων. Η μετανάστευση, η επιστροφή και η βιώσιμη επανένταξη των επιστρεφωμένων ε, των μεταναστών είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών όσον αφορά την επανεισδοχέση, εμείς ε, ε, ε, ε, θέλουμε να διασφαλιστεί μια συνεκτική και σωστή προσέγγιση που θα βασίζεται στις αρχές της εταιρικής σχέσης της αλληλεγγύης του αμοιβαίου σεβασμού των δικαιωμάτων. Στην Αφρική η μετανάστευση και η κινητικότητα έχουν θετικό πρόσημο και μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η μετανάστευση και η κινητικότητα όταν ε, αντιμετωπίζονται με σωστό τρόπο και με σωστή διαχείριση μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα και στις χώρες προέλευσης αλλά και στις ε, χώρες ε, υποδοχής. Βεβαίως ε, υπάρχουν πολλαπλά και περίπλοκα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την μετανάστευση και την κινητικότητα και επομένως ε, θα πρέπει ε, να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να αποφευθεί η παράτυπη μετανάστευση ή εμπορία ανθρώπων καθώς επίσης και η δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τους μετανάστες διάφοροι διακινητικοί κινητές. Θα πρέπει λοιπόν, ε, θεωρούμε, να διαχειριστούμε σωστά την κυκλική μετανάστευση μετά μεταξύ των δύο υπήρων. Ε, και όσον αφορά την πανδημία θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε ε, να βρεθούν ειδικέ λύσεις για την περίοδο αυτή, αλλά και γενικότερα. Ιστορικά και η Αφρική και η Ευρώπη έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ε, πανδημίας και κατά τη διάρκεια της έχει υπάρξει ειδική υποστήριξη των χωρών της Αφρικής. Κυρίες και κύριοι, ε, πρέπει να δούμε και τα ε, μακροπρόθεσμα ε, ε, στοιχεία τα οποία αφορούν την μετανάστευση και που βρίσκουν την βάση τους στην μακροχρόνια ανεργία και την δυσχερή οικονομική κατάσταση. Δυσχερή η οποία έγινε ακόμα δυσχερέστερη στην περίοδο της πανδημίας COVID. Πρέπει να δούμε την δυνατότητα ε, να ε, υπάρξει ε, σωστή εκπαίδευση έτσι ώστε να αποκτήσουν μετανάστες και εργαζόμενοι σε κινητικότητα τις δεξιότητες αυτές οι οποίες θα είναι απαραίτητες και στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρεται και την πρόσφατα εκδοθήσα δέσμη για την μετανάστευση και το άσυλο, είναι σημαντικό σημαντικό να δούμε συγκεκριμένα πεδία τα οποία ε, αποτελούν πεδία προτεραιότητας ε, και για τις ε, δύο πλευρές στο πρόγραμμα για την μετανάστευση στην Αφρική από το 2018 μέχρι το 2030 είναι σημαντικό να δούμε θέματα τράφικινγκ επί των οποίων η Επιτροπή γνωρίζουμε ότι εργάζεται αυτή τη στιγμή. Η ε, διευκόλυνση της κινητικότητας των νεαρών Αφρικανών είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα μπορεί ε, να αμβλύνει την κατάσταση που σχετίζεται με την παράτυπη μετανάστευση. Βεβαίως και η παράτυπη μετανάστευση, μετανάστες θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι χαίρουν των διαδικασιών διάσωσης και προστασίας για τους ε, νέους ε, ε, Αφρικανούς είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη η έλλειψη ευκαιριών που έχουν στις χώρες τους. Θα πρέπει να δούμε κυρίως και να σκύψουμε βοηθώντας τους νέους από περιοχές της Υπέθρου που προσπαθούν να ψάξουν καλύτερες ευκαιρίες. Επομένως, η Αφρικανική Ένωση αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναπτύξουν ιδιαίτερα προγράμματα τα οποία θα έχουν ιδιαίτερη στόχευση ακριβώς σε αυτούς τους ανθρώπους, ε, ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την ε, οικονομική ανασφάλεια ε, της γεωργίας και επομένως ακριβώς να υπάρξουν τέτοια προγράμματα που θα αναπτύξουν τις δυνατότητες των ανθρώπων αυτών στις χώρες τους. Οι δύο ήπειροι κυρίες και κύριοι θα πρέπει να να συνεργαστούν μαζί έτσι ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να διαχειριστούν σωστά ε, ε, αλλά και οι χώρες της Αφρικανικής Ένωσης να διαχειριστούν σωστά την μετανάστευση καθένα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του. Θέλουμε εναρμονισμένες ε, ε, και συνολικές κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τις αντίστοιχες κοινότητές μας στην σωστή διαχείριση της μετανάστευσης ε, και του ασύλου. Θα πρέπει επίσης να δούμε το θέμα των οικονομικών επιταγών Ε, έχουμε δημιουργήσει τρία κέντρα στην Αφρικανική Ένωση ε, και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα ε, και τα εμβάσματα και, την, ε, ε, και τις λοιπές διαδικασίες. Επίσης στο Σουδάν, στο Μαρόκο έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό κέντρο, στο Σουδάν ένα άλλο σημαντικό κέντρο. Πρόκειται για κέντρα τα οποία είναι, έχουν υψηλή επικέντρωση για θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Πιστεύουμε ότι ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε με τεχνική υποστήριξη και λυπή υποστήριξη τις χώρες οι οποίες χρειάζονται τη βοήθειά μας και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε σε μια μετανάστευση η οποία θα είναι ασφαλέστερη και η οποία θα διέπεται από κανόνες. Ε, πρέπει να σας διασφαλίσω κυρίες και κύριοι ότι υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα όσον αφορά τα θέματα αυτά από πλευρά της Αφρικανικής Ένωσης και είμαι σίγουρη ότι κάτι αντίστοιχο υπάρχει και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ολοκληρώνοντας ε, να πω ότι ε, πολλά στοιχεία βρίσκονται ε, στην Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Αφρική και βεβαίως Εκεί ε, θα πρέπει να ληφθούν ε, οι υπόψη ε, και όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την κοινωνία, την οικονομία κλπ. Πρέπει να δημιουργηθούν κοινέ ευκαιρίες, να δημιουργηθούν δυνατότητες επένδυσης και κατάρτισης κλπ. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά την σημασία ε, καλών σχέσεων μέσα από τους νόμιμες οδούς μετανάστευσης, αναγνώριση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων, ε, κοινά προγράμματα για την κινητικότητα των ε, επιστημόνων κλπ. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε την εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Θα δημιουργηθεί ένα κοινό ε, πλαίσιο που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που ε, αφορούν και συνδέονται με την μετανάστευση και το άσυλο. Η Αφρικανική Ένωση παραμένει ε, αφοσιωμένη στους στόχους αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι που μου δώσατε τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή τη διάσκεψη. Σουκρά. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Θα δώσω το λόγο τώρα, θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο στην κυρία Ούρπι Μας ακούτε? σας ακούμε κι εμείς και σας βλέπουμε. Ωραία. Αγαπητοί συμπρόεδροι, αγαπητή κυρία Επίτροπε της Αφρικανικής Ένωσης, εξοχότατοι αγαπητοί συνάδελφοι. τελεί και εμένα τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την πολύ σημαντική και επίκαιρη διακοινοβουλευτική συζήτηση για τη μετανάστευση και το άσυλο και θα ήθελα να εστιάσω στο δικό μας έργο, το πολύ σημαντικό που κάνουμε για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μόνη της να διαχειριστεί τη μετανάστευση. Χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστούμε με χώρες εταίρους επί τη βάση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και να υπάρχει ε, ε, κοινή σεβασμός από κοινού για την ευθύνη του, και ε, του καθενός. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση, την παράνομη μετανάστευση και ταυτόχρονα να βοηθηθούμε από τα ωφέλη που φέρνει η νόμιμη μετανάστευση. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν θα μείνει πίσω. Εάν η μετανάστευση τύχει σωστής διαχείρισης, μπορεί να συνεισφέρει στην κοινωνική ε, ε, στην πρόοδο της κοινωνίας και να μειώσει τις ανισότητες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η συνεργασία μας θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να αφουγκραστούμε τους εταίρους μας, να καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές τους, ποιες είναι οι ανάγκες τους και να αντιληφθούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να τους υποστήριξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η Συμφωνία για την Μετανάστευση και το Άσυλο προβλέπει την δημιουργία εταιρικών σχέσεων αμοιβαίως υποφελών ε, μεταξύ ε, με τις χώρες ε, προέλευσης και προορισμού. Εχθές είχαμε την δεύτερη συνάντηση στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νιγηρίας και συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και της κινητικότητας να βοηθήσουμε από την δική μα την πλευρά την Ιγυρία σε στόχους όπως η ισότητα των δύο φύλων, η ειρήνη και η ασφάλεια, η κοινωνική πρόνοια κτλ. Τα λέω αυτό γιατί δείχνει ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε τη μετανάστευση ε, ξεχωριστά από άλλα, από άλλα θέματα, από άλλα προβλήματα. Ε, υπάρχουν λοιπόν αυτές τις συμφωνίες, όμως χρειάζεται και η πολιτική βούληση για να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Η συνεργασία με τους εταίρους μας σε διεθνές επίπεδο πρέπει να εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Σε πολυμερές επίπεδο, στη συνεργασία με συγκεκριμένες χώρες, στην χρήση των διαφόρων πλαισίων που υπάρχουν ε, για τη μετανάστευση, όπως για παράδειγμα τις ε, διαδικασίες της Βαλέτας, της Πράγας, του Ραμπάτ κτλ. Σε αυτό το επίπεδο βλέπουμε και τη συνεργασία μας με την Αφρικανική Ένωση ως μια συνεργασία πολυμερή. Με τον ίδιο τρόπο επίσης βλέπουμε και τη συνεργασία μας με το Ενωμένα Έθνη ή με τα κράτη της περιοχής ΑΚΕ. φροντίζοντας ε, να έχουμε αυτή τη συζήτηση για τη μετανάστευση στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης που κάνουμε με τις τρίτες χώρες, μας δίνει τη δυνατότητα να, να ε, την συνδυάσουμε με θέματα όπως το εμπόριο, η δημιουργία θέσεων αναργασίας, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, ε, την εκπαίδευση και με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουμε ότι η μετανάστευση είναι και αυτή το και αυτή ένα θέμα πολιτικής κεντρικής σημασίας μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και πιο συγκεκριμένες ε, συνεργασίες όπου αυτό χρειάζεται και είναι απαραίτητο ε, για να προωθήσουμε τους στόχους μας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει πλήρης συντονισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργεί ως μια ομάδα. Όπως φάνηκε αυτό στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού, ε, χρειάζεται να υπάρχει συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Φυσικά, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράσεις που θα κάνουν τη διαφορά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα που θα τις επιτρέψουν να έχει συνεργασία και με τους διεθνείς ε, εταίρους της, κάτι που προβλέπεται και στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό ε, πλαίσιο ή επίσης το εργαλείο Ντίκη για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτες χώρες. Συνεχίζονται φυσικά, όπω γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσει στο ιστορικό τη Ένωση για το θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα τηλεσφορήσουν και ελπίζουμε ότι το εργαλείο αυτό θα μα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη συνεργασία και στα θέματα τη μετανάστευση. Σύμφωνα με την ε, πρόταση τη Επιτροπή, το 10% του εργαλείου αυτού θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων που ε, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα γενοσιουργά αιτία ε, τη μετανάστευση και δράσει διαχείριση τη μετανάστευση. Ε, η οικονομική υποστήριξη που θα προσφέρει η Ευρώπη στις τρίτες χώρες ε, θα πρέπει να βασίζεται στους στόχους πολιτικής που συμφωνούμε, αλλά βέβαια να έχει και την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ να συζητήσουμε και με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσω τις παρεμβάσει και των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σα ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τομπέ για το επόμενο μέρος της συζήτηση. Ευχαριστώ. Πριν ε, περάσουμε στον κατάλογο των συναδέλφων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, έχουμε δύο σημεία προσυζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Νίκολα Μπέι, εκπρόσωπο της, ε, του Δανέζικου Συμβουλίου Προσφύγων στην Βοσνία Ερσεγοβίνη. Για πέντε λεπτά παρακαλώ συναδέλφα έχετε το λόγο. Καλησπέρα, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Στα πλαίσια της εξωτερικής διάστασης και εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες, το Συμβούλιο μας πιστεύει ότι είναι σημαντικό ευθύ εξ αρχής να τονίσει το εξής υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξωτερική πολιτική εξαιτία του ε, αυξανόμενου προβλήματος μετανάστευση και προσφύγων μεγάλο πρόβλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και προστασίας εκ μέρους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνοντας χώρες. Ξέρουμε ότι γίνουν πάρα πολλά σε χιλιάδες ε, ε, αποστολές επιστροφής σε χώρες. Υπάρχουν ε, τεκμήρια και μαρτυρίες για προβλήματα βίας καταχρήσεων στα πλαίσια αυτών των ροών και όπως ξέρετε πρόκειται για πλήρη κατάχρηση των δικαιωμάτων τα οποία πρέπει να έχουν ετούντε άσυλο. Η πολιτική αποτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το εξωτερικό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα εξαιτία των ε, υποδομών υποδοχής του προβλήματος διαχείρισης το του γεγονότος ότι υπάρχουν όλα αυτά τα άτομα που βρίσκονται σε δινή κατάσταση που ε, αναγκάζονται να καταλύσουν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια τα οποία δεν έχουν καμία στοιχειώδη ε, ε, και δεν έχω καμία στοιχειώδη πρόσβαση στα χρειώδη. Όπω καταλαβαίνετε υπάρχει τρομερό πρόβλημα και τρομερή πίεση προ όλε τις κυβερνήσει. Το, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ σα μιλώ κυρίω για το τι έκρυβε στην Βοσνία Γεωργολτήτη. Η νέα συμφωνία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων στα Βαλκάνια. Θα πρέπει όμως όλα αυτά να γίνονται βάσει τη αρχή τη ίσης κατανομής των βαρών δεν θα ε, πρέπει να γίνονται αποτέλεσμα εκβετάλεσης όλα αυτά τα άτομα τα οποία αιτούν ε, άσυλο και πρόσφυγες. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ε, αξιοπρεπείς ε, συνθήκες ζωής και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ή ώρες με τρίτες χώρες. Η ζωρες με τριτες χωρες βοήθεια θα πρέπει να δείτε βάση ε, αντικειμενικών στόχων για την εκρίζωση της φτώχεια και για να μπορέσουν όλα τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων να εξασφαλίζονται και να έχουμε και σαφείς στόχους ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν βάσει του δικαίου να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων όποια και να είναι η θέληση κάθε χώρας χωριστά να τα εφαρμόσει. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν ειδικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις με ένα σχεδιασμό αϊφόρος και μακροπρόθεσμα στη σε εφαρμογή, ώστε να υπάρχει πρώτα απ' όλα ε, ε, πλήρη συμφωνία με τον σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και τη τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου για αυτά τα άτομα. Να σταματήσει η βία και η επιστροφή με βίο τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά σύνορα. Είναι λοιπόν πρωτορχική σημασία να υπάρχει εποπτεία στα εξωτερικά σύνορα. Θα η πρόταση να υπάρχει μία ε, σωστή ε, εποπτεία ώστε να ξέρουμε πώς γίνονται τα πράγματα στα σύνορα είναι κάτι το σωστό. Αλλά θα πρέπει να έχουμε έναν ενισχυμένο μεχανισμό για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός και κυρίως να μπορέσει να αναπτυχθεί στις περιοχές στις οποίες γίνονται αυτές οι προσπάθειες βίας ε, επιστροφής των ατόμων αυτών. Να μπορέσουμε να κάνουμε μία ε, αξιόπιστη πολιτική και τις κατάλληλες έρευνες ώστε να μπορέσει να είναι βιώσιμος αυτός ο μηχανισμός. Τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει και συμπληρωματικά ε, τρόπους προταξίας, επανένωση οικογένειας, ε, ε, προστασία όλων των μελών της οικογένειας, δυνατότητες εργασίες και να μπορέσει να εξασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες ζωής αυτών των ατόμων. Επίσης, να ενισχύσει την νόμιμη μετανάστευση και την προστασία των προσφύγων. Σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να θέσω όλα αυτά τα θέματα. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε απάντηση σε ερώτησή σας. Thank you, Mr. Bay. Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέι. Ο κύριος Μίλιμπαντ, Διευθύνων Σύμβουλος ε, της International Rescue Committee, δυστυχώς ε, δεν ε, μπορούσε να είναι μαζί μας, αλλά μας έστειλε ένα βίντεο.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 and look forward to decisive action which advances European interests and values. Thank you very much indeed. Thank you, Mr. Ο κύριος Ντομπέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μίλιμπρα για αυτό το μήνυμα μέσω βίντεο. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση ε, με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς επίσης ε, και τους βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εναλλαγή θα γίνεται μεταξύ των ομιλητών. Ένας ομιλητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα από, το, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η κυρία Μαρία Σοράγια Ροδρίγες Ράμος, η οποία είναι επικεφαλής της ε, ε, ομάδας σύνδεσης ε, με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Ροδρίγε Σοράγια. Αγαπητοί συμπρόεδροι, Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πάρω το λόγο και να συμμετάσχω βέβαια σε αυτήν την διάσκεψη ε, για την μετανάστευση και το άσυλο. Ε, ήθελα να πω ότι Οπωσδήποτε κάθε τέτοιου είδους πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πρέπει οπωσδήποτε η προσέγγιση να είναι συνολική και ολιστική και η συνεργασία να είναι μεγαλύτερη. Ε, και βεβαίως ε, για να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη και μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της Ευρώπης και των άλλων χωρών. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ε, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε το βάρος να μην πέφτει πάντα και μόνο στους ώμους των χωρών που είναι χώρες εισόδου. Ε, πρέπει να ε, ε, διασφαλίσουμε επίσης ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ήδη ευάλωτων μεταναστών. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε ότι οι μετανάστες αποτελούν ένα μεγάλο σημείο δύναμης. Το είδαμε άλλωστε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλές από τις βασικές υπηρεσίες δόθηκαν διασφαλίσεις από μετανάστες. Τρίτον, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία. Ω πρόεδρος της συνεργασία ε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου ε, ε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία για θέματα οικογένειας, ενσωμάτωσης, μετανάστευση ασύλου. Αύριο θα έχουμε μια τέτοια συνάντηση του οργάνου μας. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με τα κέντρα της Ραμπάτ και του Χαρτούμ, αλλά γενικότερα να ξέρουμε ότι μονάχα εάν συνεργαστούμε μέσα από έντονη ε, ε, και εντατική διακοινοβουλευτική συνεργασία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Τομπέ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, θα δώσω τον ε, λόγο. Δεν είναι συνδεδεμένη η συνάδελφος. Περνάμε στο επόμενο μέλο Ο κύριος Καρμέλο Μπονίτσι από το Κοινοβούλιο της Μάλτας. Δεν βλέπουμε τη σωστή εικόνα, δεν έχουμε. Περνούμε στον επόμενο. κύριος Κάρλος Σουρίνιο από το να αντιπροσωπεί με τις χώρες και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Κυρία Σουρίνιο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπορώ να συνεισφέρω στην συζήτηση αυτή της διάσκεψης υψηλού επίπεδου. Το πλαίσιο του ευρωπαϊκού Ένωση είναι το ε, καλύτερο δυνατό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε δεδομένου ότι περιλαμβάνει πολιτικές σχέσεις, δημοκρατία, συνεργασία, εμπορικές σχέσεις κτλ. Οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας όπως είπε και η Επίτροπος είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σημαντικά εξαιτία των θεμάτων τόσο σημαντικών που είναι η μετανάστευση και το άσυλο. Και πρέπει στα πλαίσια της συνεργασίας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τα θέματα της μετανάστευσης ακόμη ε, δεν έχουν επιληθεί. Υπάρχουν μεταξύ ε, των προβλημάτων ε, διαφορές και κλωσικές όσον αφορά τα θέματα ουσίας για τους μετανάστες. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε εταιρικέ χώρες με τρίτη σχέση ισχυρέ, όπω φερειπίν μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Αφρικανικών χωριών. Εμείς υποστηρίζουμε πλήρως του στόχους και τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει ισοτιμία και δεν κατορθώσουμε να επιλύσουμε τις διαφορές που υπάρχουν, ώστε να είναι επωφελής. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ των εταίρων και βεβαίως η Αφρική θέλει να εξασφαλίσει ε, όσα περισσότερα ωφέλη μπορεί για τις οικογένειες των πολιτών αυτής της ε, και υπηκών της Υπήρου που φτάνει στην Ευρώπη. Όπως είπε και συμπρόεδρος θα πρέπει για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το πρόβλημα αυτό της μετανάστευσης στην Ευρώπη, να δούμε πώς θα γίνει η δίκαια κατανομή, ώστε να μην επιβαρύνονται μόνο με άδικη κατανομή κάποιες χώρες. Στην Ευρώπη θα πρέπει να επιδείξουμε και την αλληλεγγύη μας προς όλους όσους χρήζουν προστασίας. Βάσει των αρχών του κρατικού του διεθνούς ε, ε, δικαίου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλες. Πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο να ενεργήσουμε με μία προοπτική μακροπρόθεσμη και να μην ε, ε, κάνουμε μόνο ενέργειες οι οποίες είναι κοντόφθαλμες. Θα πρέπει να ευνοήσουμε επίσης την ε, κινητικότητα, να λάβουμε υπόψη τα επανένωση των οικογενειών, τα συμφέροντα των ε, οικογενειών, άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ δυνατοί για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτά τα θέματα στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας και για τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να περιορίζετε τις παρεμβάσεις σε δύο λεπτά μόνο. Ο κύριος Καστελούτσι τώρα μέλος της Bundestag. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχεις γερμανικά, έχεις γερμανικά. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο προλεήσιος συνάδελφος καθώς με, και αυτά με τα οποία είπε η Επίτροπος. Θα πρέπει εδώ να μπορέσουμε ίσης ε, όρις να δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσει. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Και βεβαίω θα πρέπει η οικονομική ανάπτυξη να είναι σημαντική διάσταση, αλλά θα πρέπει και οι συνθήκες και οι προποθέσει να είναι καλέ. Θα πρέπει η συνεργασία μα, λοιπόν ε, για την ανάπτυξη να μην χρησιμοποιηθεί για άλλου λόγου. Θα πρέπει να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, επαναλαμβάνω, ίση όρου. Το θέμα τη μετανάστευση δεν είναι μόνο η παράτυπη μετανάστευση, η εμπορία ανθρωπίνων είναι και κάτι διαφορετικό. Και το ερώτημα που θέτω που είναι πολύ σημαντικό είναι τα άτομα τα οποία καταδιώκονται, που χρειάζονται προστασία, αυτά τα άτομα μπορούν να ε, τύχουν συνθήκων ασφαλείας. Βεβαίως μπορεί κανείς να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση, αλλά αυτή τη βασική αρχή δεν θα πρέπει να την καταστρατηγήσουμε. Έχουμε δεσμεύσεις προς αυτά τα άτομα, τις οποίες θα πρέπει να τιμήσουμε κατά προτεραιότητα. Κανένας δεν θα πρέπει να διώκεται ή να χρειαστεί να καταφύγει κάπου χωρίς να του δοθεί βοήθεια. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά. Και τρίτη παρατήρηση, όπως είπε και ο κύριος Μίλιμπαντ, η ΕΝΕΣΕΡ μας λέγει ότι θα πρέπει να έχουμε πραγματικά ε, περίπου εκατομμύριο νέες επανεγκαταστάσεις ή μετεγκαταστάσεις στα πλαίσια της πολιτικής τα επόμενα χρόνια. Δεν θα πρέπει να μιλούμε λοιπόν μόνο για μετανάστευση. Θα πρέπει να δούμε την κυκλική μετανάστευση. Θα πρέπει να δούμε την ένταξη αυτών των ατόμων στις κοινωνίες μας, τις δυνατότητες εκπαίδευσης και εργασίας κτλ. Ευχαριστώ. Of the Chamber of Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο από την Βουλή του Λουξεμβούργου στην κυρία Δεπέιν. Δεν έχει συνδεθεί, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, τότε ας προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή. Αντιπρόεδρο της πιο σημαντικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, Κυρία Άσπεργκερ, αν μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι speak. Με ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερος ευτυχής που έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα υπό την αιγίδα της Γερμανικής Προεδρίας. Και θα ήθελα να αναδείξω ορισμένα από τα θέματα σχολούν το Κοινοβούλιο. Η πρόταση που υπέβαλε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, μετανάστευση και το άσυλο είναι κατά την άποψη της πολιτικής μου ομάδας των Πρασίνων προβληματική. Ωστόσο, ως ε, σχεδόν εισηγήτρια για την στρατηγική για τις εταιρικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, έχω μια συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης αν δει κανείς την ένταξη του θέματος της μετανάστευσης τη συμφωνία μετά το Κοτονού, έχουμε δει ότι υπάρχουν διεστάμενες απόψεις, αλλά ε, τουλάχιστον ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούμε είναι ότι θα πρέπει να καταπολεμήσει κανείς τους λόγους που οδηγούν του ανθρώπους να μεταναστεύουν. Δηλαδή, να φροντίσουμε οι άνθρωποι να έχουν ασφάλεια, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, να έχουν ε, να μην λιμοκτονούν, να έχουν επίσης πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στις χώρες τους. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε και το εξή ζήτημα. Ε, μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί λόγους για να μεταναστεύουν οι άνθρωποι. Μήπως από κάποιες από τις εταιρικές της συμφωνίες ε, δημιουργούν τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν εξαγωγές που τελικά δημιουργούν προβλήματα στις ε, τοπικές ε, αγορές εργασίας, αγοράς εργασίας. Μήπως έχουμε και εμείς ευθύνες αν δίνουμε μικρά όπλα, για παράδειγμα, πουλάμε μικρά όπλα σε περιοχές του κόσμου που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι κάνουμε για την προστασία όλων αυτών των περιοχών. Πολύ συχνά όμως ξεχνάμε να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι επιζήμιες δραστηριότητες που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της αναλαμβάνουν. Επανέρχομαι σε κάτι που ακούστηκε και το πρωί, ότι η μετανάστευση μπορεί να είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί. Μπορεί να δημιουργήσουμε, μπορούμε, φροντίσουμε και υπάρξει πολιτική βούλευση να δημιουργήσουμε ε, ε ουσιαστικά διεθνή πρότυπα που τελικά θα οδηγήσουν στο να σώζουμε ζωές αντί να τις ποινικοποιούμε. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παμπίν, μέλος του, Ευρωπαϊκού, του, συγγνώμη, του Κοινοβουλίου της Σλοβενίας, υπεύθυνο για ζητήματα ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. κύριος σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρα. Είναι γνωστό ότι οι προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την πανδημία και οι προκλήσεις που το, δημιουργούν οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν υποχωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να βρει μια νέα, ε, ένα νέο βηματισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν πολλά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά όπως για παράδειγμα οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες, τις, χώρε χώρες προέλευσης. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξουν συμφωνίες, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και να συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση. Ε, εγώ συμμετείχα σε ένα συνέδριο της Europol για, την για το συντονισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και εκεί είδα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της διακίνησης δηλαδή. Επιστώνουμε επίσης ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν σταμάτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι διακινητές βρίσκουν όλο και πιο εφάνταστους νέους τρόπους να φτάνουν στην ε, Ευρώπη. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτή η κατάσταση να πάψει. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να ενισχύσουμε τις πολυμερείς συνεργασίες. πρέπει να, θα πρέπει να θέτουμε τα ζητήματα η Σλοβενία έχει και εκείνη ένα πρόγραμμα διεθνού ε, ε, αναπτυξιακής βοήθειας και πιστεύω ότι χρειάζεται να υιοθετήσουμε τα σωστά μέτρα χωρίς να ξεχνάμε την ανθρωπιστική διάσταση του προβλήματος η εξωτερική διάσταση της πολιτικής μετανάστευσης έχει άμεσες επιπτώσεις στα προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε στις χώρες μας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίζει πιο γρήγορα κρίσεις και να αξιοποιεί και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, τον κύριο Μπορέλ. Ε, έχουμε διαπιστώσει ότι η απόκρισή μας σε κρίσεις δεν είναι τόσο γρήγορη όσο πρέπει. Ελπίζω το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση να εγκριθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και να δούμε ποια εργαλεία θα δώσουμε στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν στην πράξη αυτή την ε, πιο στενή συνεργασία. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριος Καμπορ Ιβοστήρ από το Κοινοβούλιο της Κροατίας θα είναι ο τελευταίος μας ομιλητής και από ό,τι θυμάμαι ε, και παλαιό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παλαιότερα έστασε στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Έχετε το λόγο. speak button, please. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί του ομίλητη παρακαλώ. Ναι. Μπορούμε να σας δούμε και να σας ακούσουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σας από το Κοινοβούλιο της Κροατίας θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η πιο αποτελεσματική χρήση που θα μπορούσαμε να κάνουμε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής για τη διαχείριση των συνόρων. Πάρα πολλοί πόροι διατέθηκαν για την διαχείριση του ε, συνόρων για 1.200 χιλιόμετρα μεταξύ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Κροατίας. Ξέρουμε ότι έχει γίνει ένας ε, φράχτης, το ίδιο έχει γίνει και από τη μεριά της ε, Ουγγαρίας. Αντί να δαπανάμε εκεί τα λεφτά, θα πρέπει να λάβουν δεσμεύσεις οι χώρες οι οποίες θα ήθελαν να γίνουν ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουν και μέλος της Ένωσης θα μπορούσε η Frontex ενδεχομένως να βοηθήσει ώστε να μπορέσουν να χειριστούν τα σύνορά τους. Έχουν σύνορα με τη Σερβία όπως ε, ξέρουμε η Frontex επίσης αναπτύσσεται και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Θα ήταν αυτό αποτελεσματικό και θα μας βοηθούσε να ξεκονομήσουμε κάποιους πόρους που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε άλλα προβλήματα όπως Φερρυπίν το θέμα των ε, οδών διέλευσης των μεταναστών από κάποια κρίσιμα σημεία. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση σήμερα νομίζω και με το COVID ότι είναι ε, σημαντικό να ενεργούμε πάντα στα πλαίσια των κανόνων του κράτους δικαίου. Να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άλλες ε, οδοί και άλλες ροές μεταναστών, παράνομες από την Αφρική προς την Αφρική θα πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια της συνεργασίας κάτι θα πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας λοιπόν και να δώσουμε τους πόρους που χρειάζεται για να είναι πιο αποτελεσματική λύση των προβλημάτων εκεί που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ, ε, η επίτροπο κυρία Ουρπιλάιν έπρεπε να φύγει. Έχει μια άλλη συνεδρίαση. Όμως θα ήθελα να πω εξ ονόματος ε, της ε, Προεδρίας, μια και είμαι συμπροέδρος, να ευχαριστήσω λοιπόν ε, για την συνεργασία και για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία κάνετε και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλετε στη συζήτησή μας. Θα ήθελα τώρα ξανά να δώσω τον λόγο στην συμπρόεδρο Μόνικα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκρεγόρτσιτς. Θα προχωρήσουμε τώρα με το δεύτερο τμήμα της συζήτησής μας. Εξ αρχής θα ήθελα να σας ζητήσω αγαπητοί συνάδελφοι να σέβεστε τον χρόνο που σας έχει δοθεί είναι δύο λεπτά. Τώρα θα δώσω τον ε, λόγο ε, από την πλευρά της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κυρία Βίσελερ Λίμα. Καλό απόγευμα, λέει η κυρία Βίσελερ. Ο τίτλος ε, του πάνελ μας βρίσκεται ακριβώς εις τα μελήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν διαλέγει μια, όταν διαλέγει μια οικογένεια να πάει σε μια άλλη χώρα, αυτό δεν ε, αποτελεί πρόβλημα. Τα μαζικά, οι μαζικές μετακινήσεις είναι αυτές οι οποίες ε, προκαλούν τον ε, φόβο και δεν μπορεί κανείς να, αγνωρίσει, να αγνοήσει τους φόβους αυτούς, έστω και αν είναι αβάσιμοι γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην ε, κοινωνία. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν, κάνουν μια επιλογή ε, και αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να βοηθήσουν οι εταιρικές σχέσεις και αυτές οι συνολικές εταιρικές σχέσεις είναι αυτές οι οποίες μπορούν να αλλάξουν και τις συνθήκες διαβίωσης επιτόπου Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, πραγματικά θέλουν να μείνουν στις χώρες τους ε, και μια αναπτυξιακή πολιτική η οποία θα τους δίνει το δικαίωμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την Αφρική πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και θέλω κατά την έννοια αυτή και εντός του πλησίου της συζήτησής μας να πω ότι η σχέση αυτή θα πρέπει να είναι σχέση μεταξύ ισοτήμων όπου ο καθένας από τους δύο ισότιμες ε, ε, ε, εταίρους προσπαθεί να προωθήσει τα δικά του θέματα σε σεβασμό όμως του άλλου. θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, χώρες από τις οποίες ξεκινούν οι μετανάστες έτσι ώστε να μην ε, υπάρχει διαρροή εγκεφάλων συστηματική η οποία τελικά ε, θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στις χώρες εκκίνησης. Θα πρέπει ε, λοιπόν ε, ισότιμες σχέσεις ε, και ισότιμα να αντιμετωπίζονται και οι δύο χώρες. Επίσης, οι δύο πλευρές μάλλον. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές, δεν μπορεί να υπάρχει ισότιμη σχέση εάν από τη μία πλευρά υπάρχει παρίσφρηση στα εσωτερικά της άλλης χώρας ή από την μία πλευρά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται βία, οι οποίοι διώκονται. Ευχαριστώ πολύ. Πέντρο Φελίπε Σοάρες από την Πορτογαλία. Από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο είναι ο επόμενος ομιλητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Πορτογαλικής Βουλής. Δυστυχώς ε, δεν είναι συνδεδεμένος ο κύριος Σοάρες. Να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια επομένως. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπετίνα Βόλακ. Από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο λέει η κυρία Βόλατε, Ευχαριστώ πολύ και για ε, όλα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσε όλες οι παρεμβάσει. Υπόθηκε και προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με τις τρίτες χώρες και μάλιστα μέσα σε πλαίσια διαφάνειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε φορά θα πρέπει να ελέγχεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε εταιρική σχέση, αλλά αυτό δεν γίνεται συστηματικά Σκέφτομαι ας πούμε την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ε, την ε, κατάσταση στην ε, χώρα αυτή και δεν μπορεί κανείς να υποκριθεί ή να καμωθεί ότι δεν γνωρίζει τι γίνεται, τι συμβαίνει επί τόπου. Ε, απ' την άλλη πλευρά εξωτερικοποιούμε την πολιτική ασύλου που στην ουσία σημαίνει ότι εμείς εξωτερικοποιούμε οποιαδήποτε ε, ευθύνη ενώ η κατάσταση επιτόπου και η γνώση που έχουμε για την κατάσταση επιτρόπου είναι τρομερή. Πότε θα διαλευκανθούν αυτά, πότε θα τα καταλάβει η Κομισιόν, πότε θα τα λάβει η υπόψη της. Δεν είναι δυνατόν ε, εφημερίδες όπως η Σπίγκελ ας πούμε να αναλαμβάνουν, να ξεκαθαρίσουν το τοπίο ή να καταγγείλουν την κατάσταση. Ε, βεβαίως τα θέματα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά, επαναλαμβάνω, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε τους διάσταση. Γνωρίζετε τον προβληματισμό που έχουμε, κυρίως ε, όσον αφορά ας πούμε σχέσεις με χώρες όπως η Τουρκία ή το Αφγανιστάν. Θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε συνεκτική προσέγγιση ε, με βάση μια πραγματική και ουσιαστική προστασία. Ε, και κυρίως να μην λησμονούμε τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού και πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Άγγελος Συρίγος ε, από την Ελληνική Βουλή. Παρακαλώ κύριε Συρίγο έχετε το λόγο. ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ γενικότερα που μας δίνετε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον τόσο σημαντικό διάλογο για ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Για περισσότερα από 13 χρόνια, τρεις συγκεκριμένες χώρες παραμένουν στην κορφή των εισόδων ε, προσφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία οι αριθμοί εισόδου μπορεί να αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο. Τη μία χρονιά προηγείται η Ελλάδα, την άλλη η Ιταλία ή η Ισπανία. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι από την ένταξη των νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το 2004, οι τρεις συγκεκριμένες χώρες παραμένουν πάντοτε στο επίκεντρο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Για εμάς λοιπόν η συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι απαραίτητη. Η αρχή more for more για τις χώρες που συνεργάζονται και less for less για τις χώρες που δεν δέχονται να συνεργαστούν είναι απαραίτητη για τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι προφανές ότι η πίεση πρέπει να είναι ενιαία και συντονισμένη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να λειτουργήσει ένας κοινό ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών. Μόνον μέσα από ένα τέτοιο σχήμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πολλαπλασιάσει τη δυνατότητα πιέσεων και θα προσφέρει βοήθεια προς τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Και εμείς ευχαριστούμε. Δέτλερ Ζάεφ, ο επόμενος ε, ομιλητής από το Bundestag, Γερμανική Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου διατυπώνεται σε πέντε νομοθετήματα και τέσσερα κανόνες χωρίς ε, νομοθετική στάτους. Όλα αυτά φαίνονται πολύ καλά φτιαγμένα στα χαρτιά, ωστόσο δεν καταφέρνουμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. παράδειγμα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα δημιουργήσει το Task Force, την, την ομάδα εργασίας η οποία προβλεπόταν για την ε, εφαρμογή του κοινού συστήματος ασύλου. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχουν ήδη ε, συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ κρατών, ε, μεταξύ κρατών της Ένωσης και τρίτων χωρών. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η εξωτερική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες θα πρέπει να συνεργαστούν επιτέλους οι διάφοροι αρμόδιοι επίτροποι και διάφορε γενικές διευθύνσεις τους, έτσι ώστε να καταλήξουν σε μια σωστή περιγραφή πλήρη της κατάστασης, έτσι ώστε να μπορέσουμε τελικά να συνεργαστούμε και να εφαρμόσουμε τη λεγόμενη εξωτερική διάσταση της πολιτικής ασύλου. Θα δώσω τώρα το λόγο, λέει η κυρία ε, Γκρεκότση, στον κύριο Ζήμιοκ, την ε, Επιτροπή ανάπτυξη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ δυστυχώς. Και σήμερα έχω την αίσθηση ότι αναμασούμε τη, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, ε, πάντοτε έχουμε μία ε, αναφορά στη σημασία που έχουν οι εταιρικέ σχέσεις με τρίτες χώρες, πάντοτε έχουμε και μία συναισθηματική αν θέλετε προσέγγιση, όμως ε, κατά την άποψή μου χρειάζεται μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Δεν άκουσα τίποτα για παράδειγμα για την αιρεσιμότητα, δηλαδή ότι θα πρέπει να τεθούν ε, ενώπιον των ευθυνών τους οι χώρες προέλευσης. Δηλαδή, όταν έχουμε μια χώρα που το 1 τρίτο του ΑΕΠ της προέρχεται από δωρεές και από αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάει να πει ότι κάτι δεν έχει λειτουργήσει καλά εάν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται επί πολλά χρόνια. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες μας. Είναι προφανές ότι μπορεί να υπάρχουν διεθνείς ευθύνες, αλλά αυτές δεν συμπεριλαμβάνουν και την ε, το να, φροντίσει κανείς το πληθυσμό σε όλες τις τρίτες χώρες. Ε, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε μετανάστες που το επιθυμούν, λέμε, να επιστρέψουν στην χώρα τους. Όμως αυτό κατά την άποψή μου είναι αφελές. Θα είναι πολύ δαπανηρό να επιστρέψει κάποιος στην Αφρική και τελικά θέτω και ένα ηθικό ερώτημα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Ε, είναι γνωστό ότι κραπανούμε πολλά χρήματα για μελέτες. Η κυρία Φοντερ Λάιεν είναι ιδιαίτερος ε, επιρρεπής σε τέτοιου είδους δαπάνες. Όμως τελικά κάνουμε και κάποιες μελέτες που να μας δείχνουν εάν οι πολιτικές μας είναι ε, εφαρμόσιμες ε, ή απλώς έχουμε μια τοπική προσέγγιση που θα προ... τέριαζε περισσότερο στην Άστερ Λίντρικεν. Ε, θέλω λοιπόν να ξαναδούμε γενικότερα το μοντέλο με το οποίο πορευόμαστε. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, κυρία Πούρα από το ε, Φινλανδικό Κοινοβούλιο, Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσια Διοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που παίρνω το λόγο αμέσως μετά τον ομιλητή που προηγήθηκε. Γιατί πιστεύω πως είναι σημαντικό να συζητήσουμε και το θέμα των επιστροφών. Ένα θέμα για το οποίο δεν ε, συζητήσαμε αρκετά ακόμα. Κατά την άποψή μου όλο αυτό το σύστημα για τις επιστροφές θα πρέπει να βελτιωθεί. Θα πρέπει να δούμε τελικά ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την επιστροφή ανθρώπων στις χώρες προελεύσευσής τους ε, και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες, μεγαλύτερος αριθμός ε, αφήξεων μεταναστών είναι προς την Ευρώπη. Ε, ανεξαρτήτως του εάν αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται ή όχι διεθνούς προστασίας. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένας πόλος έλξης στην Ευρώπη και σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται αδύνατο να διαχειριστεί κανείς το φαινόμενο. Και το, το ζήτημα αυτό, το πρόβλημα αυτό επηρεάζει και άλλους τομείς πολιτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να έχουμε σαφείς και αυστηρές προδιαγραφές ερεσιμότητας σε, στην πολιτική ε, της αναπτυξιακή συνεργασία και στην πολιτική του διεθνού εμπορίου που έχουμε με τρίτε χώρε. Πιστεύω ότι αυτό το εργαλείο δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει επαρκώ. Ε, δεν θα είμαστε σε θέση εμείς από την Ευρώπη να λύσουμε τα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Μισελ Γιάκτσιτς, τώρα, πρόεδρος της ε, Επιτροπής Δικαιοσύνης του Κροατικού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω, λέει η Πρόεδρος, να τηρείτε το όριο των δύο λεπτών στις παρεμβάσεις σας για να μπορέσουν να πάρουν το λόγο όλοι όσοι το επιθυμούν. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, but Mr. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος είπε ότι θέλαμε να πούμε εκ μέρους του Κοινοβουλίου της Κροατίας δεν θέλω να αφαιρέσω χρόνο από τους άλλους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Μόνικα Γονσάλε, μέλος τη Επιτροπής ανάπτυξη. Προς το παρόν δεν είναι συνδεδεμένη. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Ρουί Σίλβα, μέλος της ε, Πορτογαλικής, ε, ε, του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου μέλος της Επιτροπής Άμυνας. Δεν είναι συνδεδεμένος. Τελευταίος. Στην λίστα μου, ο Μουνίρ Σατουρί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέλος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Από τη δεκαετία του 80 ξέρουμε ότι άλλαξαν τα πράγματα στα θέματα συνεργασίες και πολλές ε, φορές ε, ε, με τη συνεργασία και τρίτων χωρών πολλά πράγματα έχασαν την ισορροπία τους. Νομίζω ότι όλοι έχουν υπογράψει την ε, συμφωνία στην ε, θεωρία, αλλά πρέπει να πω ότι οι πολιτικές μετανάστες νομίζω ότι έχουν γίνει πολλές ε, φορές με κατασταλτικές πολιτικές. Οι γείτονες πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα της υπεργολαβίας σε θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπως μας δείχνει η Λιβύη και η Τουρκία υπάρχουν προβλήματα πολλά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες διακριτικές και υπόγειες συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν και πολλές φορές ε, μας εμποδίζει αυτό από το να κάνουμε εμείς ελέγχους. Θα πρέπει να κάνουμε διάφορες ερευνητικές επιστολές και να υπάρχει διαφάνεια γιατί ό,τι ακριβώς γίνεται στη Μεσόγειο κυρίως για να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Θα πρέπει επίσης σε αυτά τα θέματα να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες των σχετικών οργανισμών. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ε, ε, διάφορες ε, ΜΚΟ και τους οργανισμούς οι οποίες σέβονται τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα διότι υπάρχουν κάποια πολλά προβλήματα. Θα πρέπει να κάνουμε έκκληση ώστε να μπορέσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική μεταναστευτική βάση των ατόμων και όχι των πολιτικών θεωρητικά. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα στον ε, Πίτροπο Σαμίρα Ελφαντήλ για μια σύντομη παρατήρηση και συνεισφορά στις συζητήσεις που έχουμε. Κυρία Επίτροπε, είστε συνδεδεμένοι. Ε, θα έρθουμε σε επαφή μαζί της. Δεν είναι συνδεδεμένη, διότι μας είχε πει ότι στις 3.30 θα αποσυνδεόταν. Έχουμε αργήσει λίγο συζήτηση, όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις ε, παρατηρήσεις. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ καρποφόρος και σημαντική συνεισφορά στην ε, κοινοβουλευτική διπλωματία, τη δική μας και όλων των χωρών. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με σωστό τρόπο σε όλη τις προκλήσεις για θέματα μετανάστευσης με τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Είμαι πεπισμένη ότι θα γίνουν και άλλες παρεμφερείς συνεδριάσεις ε, για τις επόμενες προεδρίες, Πορτογαλική για τις επόμενες. Κύριε Τομπέ, χαίρομαι και Αισθάνθηκα μεγάλη τιμή που σήμερα μπόρεσα μαζί σας να συμπροεδρεύσω. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω και πάλι το λόγο για να καταλήξετε κι εσείς τα συμπεράσματα της συνεδρίασης αυτής. Ευχαριστώ, Μόνικα. Ευχαριστώ πολύ, Μόνικα φτάνουμε στα συμπεράσματα και θα ήθελα να δώσω το λόγο πριν ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας σε δύο συναδέλφους. Πρώτο, στον κύριο ε, Μπέι, αν θέλει να αντιδράσει σε κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν από τους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Δύο λεπτά, σε δύο λεπτά να μας τα πείτε, αν είναι δυνατόν, κύριε Μπέι. Ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά που μου δίνετε το λόγο. Ακούσαμε πολλά για ολιστική προσέγγιση και διαχείριση της μετανάστευσης. Εγώ νομίζω ότι επί της ουσίας δεν πρέπει απλώς ε, να αποτρέψουμε την ε, άφηξη νέων μεταναστών, αλλά την προστασία των ανθρώπων αυτών. Οι κανόνες της διεθνούς προστασίας ε, θα πρέπει να αυξηθεί. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια πιο στοχευμένη εταιρική σχέση βεβαίως ε, με όμως προϋπόθεση την αμοιβαία συμμόρφωση προς τις αρχές των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ λίγο, κύριο κύριος Τομπέ και τώρα θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής Ντρουά, την κυρία Μαρία Ρενά. Μαρία, έχεις ε, τον λόγο έτσι ώστε να ολοκληρώσεις ε, ε, συμπερασματικά την συζήτησή μας. Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τομπέ, ευχαριστώ πολύ και όλους όσοι πήραν τον λόγο, κυρίως δε ευχαριστώ τους καλεσμένους μας ε, που, μας, που έριξαν άπλετο φως ε, στα θέματα της μετανάστευσης. Αυτή τη στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι επιθυμούν αλλά και υποχρεούνται να μεταναστεύσουν λόγω της πολιτικής αστάθειας, λόγω της κλιματικής αλλαγής ε, και από άλλους λόγους. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που μεταναστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση. 90% των μετακινήσεων ε, γίνονται μέσα στην ίδια Ήπειρο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τα ε, συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Ε, η ε, ομιλήτρια ε, η κυρία Μίρα Ελφαντήλ τα ανέφερε τα θέματα αυτά. Μιλάμε για μια αφρικανική πραγματικότητα η οποία είναι δυσχερής. Επίσης θα πρέπει η εταιρική σχέση να είναι βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και να είναι σχέση μεταξύ ομοτήμων. Η Επίτροπος κυρία Γιούτα Ουρπιλάινεν είπε ότι η εταιρική σχέση θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη διαφορετικά θα είναι ανεπιτυχής. Κανείς δεν είναι κατά της συνεργασίας. Όλοι θέλουν την συνεργασία αυτή, αλλά θα πρέπει να είναι συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Το Refugee Council ε, βασίζει την προσέγγιση του ε, ε, στον σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, όλων των μεταναστών. Είναι παράνομες οι επαναπροωθήσεις και αντιτίθεται στην αρχή ε, του non-refoulement και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε με μακροχρόνια και στοχευμένη χρηματοδότηση τις χώρες έτσι ώστε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, όλοι σχεδόν πλην δύο ε, οι παρεμβαίνοντες ε, αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών. Ε, διότι όλη αυτή η κατάσταση αφορά και έχει αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν όντως να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Κανείς από τους ε, παρεμβαίνοντες ε, δεν ε, αναφέρθηκε σε συνεργασία υπό όρους. Όμως αναφέρθηκε από πολλούς ο μηχανισμός προϋποθέσεων βασισμένος στην, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπε και η πρόεδρος Βοντερ Λάγεν, μετανάστευση υπάρχει από τις αρχές της ανθρωπότητας. Αυτή πλέον θα πρέπει να γίνεται βάσει των καθολικών ανθρωπιστικών αρχών και των αξιών επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει των αρχών των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει λοιπόν το κατάλληλο πλαίσιο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση μιας σωστής και κατάλληλης για τον 21ο αιώνα πολιτικής μετανάστευσης σε Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ευχαριστώ και την ε, συμπροεδρό μου Μόνικα Γκριγκόρτσιτς. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι πήραν τον ε, λόγο από τις χώρες τους ε, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ όλους για αυτήν τη στρογγυλή τράπεζα. Σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει η καταληκτική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε.